Οι καλές σχέσεις με την Παλαιστίνη για μας την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μεγάλη σημασία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο πιο σημαντικός εταίρος της Παλαιστίνης στις χρηματοοικονομικές, οικονομικές και ανθρωπιστικές ε, σχέσεις. Μια ε, Παλαιστίνη που να λειτουργεί σωστά είναι και ηθικό καθήκον για μας. Κύριε Πρόεδρε Αμπάς, αφιερωθήκατε, αφιερώσατε τη ζωή σας στο Παλαιστινιακό στην αναγνώριση της Παλαιστίνης, στην ελευθερία και χωρίς βία. Ήσασταν από τους αρχιτέκτονες της Ειρηνευτικής Διάσκεψης Μαδρίτης και της Συμφωνίας του Όσλο. Μέχρι σήμερα αποτελείται ορόσημο της Ειρηνευτικής Διαδικασίας στη Μέση Ανατολή. Σήμερα η παρουσία σας εδώ, μετά την ομιλία του Ισραηλινού Προέδρου Ρίβλιν, χτες, είναι ένα ισχυρό μήνυμα ότι η βούληση για μια αηφόρο και βιώσιμη ειρήνη μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης παραμένει ζωντανή. Σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να εξάρω την ε, ακούραστη εργασία της κυρίας Μογκερίνη, η πάτης εκπροσώπου που παρευρίσκεται σήμερα το πρωί, όπως ήταν παρούσα και χτες το απόγευμα. Καλώς ορίσατε και εσείς κυρία Μογκερίνη. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Σεπτέμβριο 2015 απεφάθη για ε, μία λύση δύο κρατών βάσει των συνόρων του 1967 με ε, την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα και των δύο κρατών. Σε αυτή τη λύση των δύο κρατών θα πρέπει να υπάρχει ένα Ισραήλ που να ζει με ασφάλεια, το είπα και χτες και το υπογράμμισα, αλλά και μια ανεξάρτητη, δημοκρατική, ε, ε, ζωντανή Παλαιστίνη που να είναι ένα κράτος βιώσιμο με συνοχή και θέλω να το υπογραμμίσω και σήμερα. Και θα πρέπει να ζουν με ασφάλεια χέρι με χέρι, δίπλα-δίπλα. Για να γίνει αυτό χρειάζεται πρώτα να τερματιστεί η βία. Κανένας πολιτικός στόχος δεν δικαιολογεί το τυφλό μίσο την υποδάβλησή του ή το, την τρομοκρατία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδικάζει και όχι για πρώτη φορά ε, την επέκταση των Ισραηλινών επικισμών καθώς επίσης ε, και την εκτόξευση ρουκετών προς το Ισραήλ από ομάδες ε, μαχητών. Αυτό οδήγησε σε έναν αποκλεισμό της Γάζας που θα πρέπει να λυθεί και το έχουμε ζητήσει και έχουμε ζητήσει και μια συμφιλίωση. Συμφιλίωση μεταξύ των Παλαιστινίων για ε, συγγνώμη, για συνέστηση, ενσυναίσθηση και μεταξύ των Παλαιστινίων αλλά και μεταξύ Πανεστινίων και Ισραηλινών. Αυτό είναι αναπόσπαστο στοιχείο της ενευτικής διαδικασίας για την οποία εσείς αγωνίζεστε. Σας καλωσορίζω και ονόματος όλων των συναδέλφων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και σας δίνω αμέσως με χαρά το λόγο. Παρακαλώ. بسم الله Κύριε Πρόεδρε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κύριε Σούλτς, κυρίες και κύριοι βουλευτές, πρώτα πρώτα, επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω για αυτή την πρόσκληση να έρθω να απευθυνθώ σε εσά εδώ στο ημικύκλιο γιατί τρέφω θαυμασμό για το δημοκρατικό μοντέλο το οποίο έχετε οικοδομήσει μέσα σε αυτή την πολυμορφία γλωσσών και πολιτισμών. Πρόκειται για καθρέφτη που αντιστοιχεί στον υψηλό πολιτισμό και στις ευγενείς ανθρωπιστικές αρχές που εκπροσωπούν οι λαοί σας, οπότε τρέφω σεβασμό και σας ευχαριστώ για τις θέσεις που έχετε υιοθετήσει για τις τοποθετήσεις σας όσον αφορά την αποκατάσταση της ειρήνης και της δικαιοσύνης στην πατρίδα μου την Παλαιστίνη. Και επιτρέψτε μου να σας μεταφέρω τους χαιρετισμού του λαού μας που προσβλέπει στο κοινοβούλιο σας. Και Δι' αυτού, επίσης, παρακολουθούμε το έργο των επιμέρους κοινοβουλευτικών επιτροπών. Θεωρούμε ότι είστε στήριγμα για την ελευθερία και ανεξαρτησία μας. Σας ευχαριστούμε για κάθε μορφή βοήθειας που μας έχετε χορηγήσει. Έτσι Νομίζω ότι θα μπορέσουμε και εμείς να οικοδομήσουμε τα θεσμικά όργανα του κράτους μας και έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε ένα δημοκρατικό καθεστώς που διακρίνεται από υπευθυνότητα και σεβασμό των διεθνώς ισχυόντων κριτηρίων για ένα κράτος δικαίου που διαπνέεται από σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν μπορώ παρά να τιμώ το κοινοβούλιο σας, αλλά και τις συστάσεις που έχετε απευθύνει σε διάφορες ε, χώρες που ε, στη συνέχεια αναγνωρίζουν την Παλαιστινιακή Αρχή. Όλα τα κοινοβούλια θέλω να ευχαριστήσω που με τη σειρά τους συστήνουν στις κυβερνήσεις τους να αναγνωρίσουν το Παλαιστινιακό κράτος. Όταν μιλούμε για τη λύση των δύο κρατών, θα πρέπει τα δύο κράτη να είναι ανεγνωρισμένα και όχι μόνο ένα από τα δύο κράτη. Κυρίες και κύριοι, από το 1917 από τον Παλφούρ έχουν περάσει 100 χρόνια. Από την Άκμπα, από την καταστροφή που μας χτύπησε και το 1948 είχαμε δεχθεί επίθεση από τον Ισραηλινό στρατό που προέβη σε σφαγιασμό του λαού μας και γι' αυτό και είχαμε εκατοντάδες χιλιάδων ε, συμπατριωτών μας οι οποίοι ζούσαν ειρηνικά και αναγκάστηκαν να εκτοπιστούν. Περισσότερα από 480 χωριά σβήστηκαν από το χάρτη. Εκεί ο λαός ζούσε ειρηνικά επί χιλιάδες ετών. Το 67 κυρίες και κύριοι το Ισραήλ κατέλαβε την Ανατολική Ιερουσαλήμ την Υπεριορτανία και τη Γάζα. Οπότε και χιλιάδες Παλαιστινίων αναγκάστηκαν να εκτοπιστούν σε Επιρδανία και Γάζα. Το ελάχιστο μπορεί να πει κανείς όταν αντικρίζει αυτό το τοπίο είναι το ότι η Παλαιστίνη ως χώρα και ως λαός έχει μια ιστορία, μια ταυτότητα, μια κληρονομιά. Πρόκειται για μια γεωπολιτική ταυτότητα που έχουμε και έχει δεχθεί το χτύπημα ιστορικής σφαγής και κατοχής που δεν έχει προηγούμενο στον 20ο αιώνα. Τώρα βέβαια βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα και όλα αυτά υπό τα βλέμματα της διεθνούς κοινότητος και των ηγετιδών δυνάμεων. Κυρίες και κύριοι, περάσαμε από μαύρες σελίδες στην ιστορία μας και ακόμα βρισκόμαστε σε τέτοια κατάσταση γιατί ο λαός υποφέρει στην ίδια του την πατρίδα από κατοχή και καταπίεση. Πρόκειται για αυθαιρεσία, πρόκειται για ρασισμό, απεχθή. Ζούμε ως πρόσφυγες μέσα σε ένα περιβάλλον δύσκολο και θα πρέπει να αντισταθούμε για να μείνουμε στην ίδια μας την πατρίδα. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπαθίες μας, ώστε να τεθεί ένα τέρμα σε αυτή την κατοχή. Να προσπαθήσουμε μέσω ε, πολιτικής, μέσω της διπλωματικής οδού και της ειρηνικής οδού. Και προχωρήσαμε σε διεθνές επίπεδο και καταβάλουμε αυτές τις προσπάθειες. Όμως δεν σημειώνεται πρόοδος όσον αφορά τις σχέσεις με το Ισραήλ. Εμείς δεν φιδόμεθα προσπαθειών, ώστε να υλοποιούμε τις συμφωνίες που συνάπτονται και τιμούμε τις δεσμεύσεις μας και θέλουμε και η άλλη πλευρά να κάνει το ίδιο. Όμως το Ισραήλ αρνείται ακόμα και τις ίδιες τις υποσχέσεις του να τηρήσει. Και συνεχίζεται η καταστολή και αυτού του είδους η ηγεμονική πολιτική σε όλους τους τομείς του βίου. Εμείς βλέπουμε το Ζαήλ να προσπαθεί να αλλάξει την πραγματικότητα στην ε, Ιερουσαλήμ. Προσπαθεί να αλλοιώσει την ιστορική ταυτότητα της πόλης. Και επίσης ε, επιτίθενται και καταστρέφουν τόπους λατρείας χριστιανών και μουσουλμάνων. Πρόκειται για απεικιοκρατική πολιτική, συνεχίζονται οι απαλωτριώσεις, ε, ακινήτων, γης και καταστροφές ε, σπιτιών, φυλακίσεις χιλιάδων Παλαιστινίων. Σήμερα δε η βία διαπνέει όλους τους τομείς της ε, ζωής μας και υπάρχει παντού πνεύμα εξτρεμιστικό. Βλέπουμε τους έπικους τους Ισραηλινούς οι οποίοι έχουν κάψει σπίτια όπως την οικογένεια Κάψα ε, και με αυτούς τους εμπρισμούς υπάρχουν και νεκροί. Κάθε μέρα ε, έχουμε άσκηση βίας, έχουμε εκτελέσεις χωρίς δίκη και πρόκειται για μια πολιτική, για μια ε, πολιτική που έχει προσφυγεί του Ισραηλινούς. Ήδη από το εσωτερικό του Ισραήλ υπάρχει επίκριση στην κυβέρνηση. Ο κύριος Χέρτζοκο, Γιαλόμ, ε, και ο Γεχούντ Μπαράκ. Πολιτικοί με ξέχουσε θέσεις στο παρελθόν και όλοι αυτοί αλλά και πάρα πολλοί δημοσιογράφοι οι οποίοι ισχυρίζονται ότι η σημερινή συμπεριφορά του Ισραήλ είναι φασιστική και ρατσιστική ακριβώς έτσι χαρακτηρίζουν την πολιτική του Ισραήλ. Έχουμε το ψήφισμα 181 του ΟΗΕ και έχουμε τότε το κόψιμο στα δύο της ε, Παλαιστίνης. Σχεδόν μισό-μισό. Όμως 87% της επικράτειας η 78% διορθώνει το 48% το κατέλαβαν οι Παλαιστίνοι δια των όπλων αυτό έκανε οι Παλαισ... και στη συνέχεια είχαμε και τον πόλεμο το 67 ακόμη αναφέρονται πολλοί σε αυτό το ψήφισμα αυτό το ψήφισμα λένε δεν θα έπρεπε να λαμβάνεται υπόψη ολόκληρο αλλά μόνο ορισμένα χωρία αυτού του κειμένου. Εγώ όμως θεωρώ ότι θα πρέπει το ψήφισμα αυτό να ισχύει 100% και παρά όλων αυτών των ψήφισμάτων, αποφάσεων της διεθνούς κοινότητα και των προσπαθειών υπέρ του να υπάρξει μια λύση δύο κρατών ακόμη δεν απολάβουμε ανεξαρτησία ως κράτος παρά το ότι είμαστε κράτος μέλος του ΟΗΕ από το 2012. Και επίσης έχουμε προσχωρήσει σε διάφορους διεθνούς οργανισμούς και έχουμε προσυπογράψει διάφορες διεθνείς συνθήκες και 138 χώρες μας έχουν αναγνωρίσει. Παρ' όλα αυτά και για να προχωρήσουμε προς την ειρήνη Επιθυμούμε να τερματιστεί ε, αυτή η περίοδος ετών ολόκληρων ε, δεινών ε, και αγώνων, δεχτήκαμε να δημιουργηθεί το Παλαιστινιακό κράτος σε επικράτεια μικρότερη του 25% των ιστορικών εδαφών. Δεχτήκαμε να δημιουργηθεί στο 22% εντός των συνόρων του 1967. Παρά τη μεγάλη αυτή θυσία, από τη διάσκεψη της Μαδρίτης και μετά και από τις συμφωνίες του Όσλο και μετά δεν έχουμε προχωρήσει καθόλου. Ε, έχει αποτελματωθεί η διαπραγμάτευση. Διαπραγματευόμαστε για τη διαπραγμάτευση, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Αυτό μας επιβάλλει το Ισραήλ που προσπαθεί να κερδίσει χρόνο έτσι ώστε να αλλάξει την πραγματικότητα επιτόπου, να ε, δημιουργήσει τετελεσμένα έτσι ώστε να απομακρυνθεί η λύση των δύο κρατών. Σήμερα το Ισραήλ συνεχίζει την πολιτική επικισμού, συνεχίζει να μας ε, απαλωτριώνει ε, τις γέες μας και να χτίζει αυτό το ρατσιστικό τείχος. Υπάρχουν πολλά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που έχουν ζητήσει από το Ισραήλ να σταματήσει τον επικισμό που ζητούν να εκριζώσει αυτό το φαινόμενο. Παρ' όλα αυτά το Ισραήλ εξακολουθεί σε αυτή την τακτική. Συνεχίζει τα έργα επικισμού και εμείς απαιτούμε από το Ισραήλ να παγώσουν όλα αυτά, να παγώσουν ε, οι διαδικασίες και ο επικισμός για να αρχίσουν οι διαπραγματεύσεις. Ούτε καν αυτό δέχεται το Ισραήλ να παγώσει ε, ο επικισμός. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι το Ισραήλ κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι ετών έχει ε, ξεκινήσει τρεις πολέμους στη ε, Γάζα, ε, σκοτώνοντας χιλιάδες ανθρώπους. Και δεκάδες παλαιστινιακές οικογένειες. Δεκάδες, εκατοντάδες οικογένειες έχουν εξαφανιστεί. Έχουν χαθεί από το ληξιαρχείο από το δημοτολόγιο. Εξαφανίστηκαν. Αφανίστηκαν μετά τους τρεις πολέμους που εξαπέλυσε το Ισραήλ στη Γάζα. Έχει καταστρέψει ε, ε, έχουν καταστρέψει και εργοστάσια ε, και υποδομές και ένα εκατομμύριο Παλαιστινίων φυλακίστηκαν από τότε που άρχισε η κατοχή. και ακόμα έχουμε 7.000 εχμαλώτους πολέμου. Άλλο ε, θέμα λοιπόν, απέναντι σε αυτή την επικίνδυνη και πικρή πραγματικότητα. Αναρωτιέμαι, μήπως έχει έρθει η ώρα να τερματιστεί κυρίες και κύριοι Ισραηλινή κατοχή της Παλαιστίνης. Γιατί δεν εφαρμόζεται το διεθνές δίκαιο. Για ποιο λόγο το διεθνές δίκαιο δεν εφαρμόζεται στο Ισραήλ. Όταν ένα κράτος επιτίθεται σε ένα άλλο, εξεγείρεται ο κόσμος όλος ως ένας άνθρωπος για να τιμωρήσει τον εισβολέα, εκτός από το Ισραήλ, το οποίο δικαιούται να μας ε, επιτίθεται ατιμωρητή. Για ποιο λόγο ε, τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών παραμένουν κενό γράμμα όταν πρόκειται για την Παλαιστίνη και για τα δικαιώματα του Παλαιστινιακού λαού. Μέχρι πότε το Ισραήλ θα απολαμβάνει αυτή την ατιμορρησία του και θα αρνείται την ειρήνη. Μέχρι πότε θα αναγνωρίζεται η η ιστορική ε, αδικία που υφίσταται ο Παλαιστινιακός λαός. Κυρίες και κύριοι, ο λαός μας θέλει να ζήσει σε συνθήκες ελευθερίας, αξιοπρέπειας, ε, στην επικράτειά του, όπως κάθε λαός σε αυτόν τον κόσμο. Ο λαός μας δεν πρόκειται να δεχθεί τη συνέχιση της κατοχής και του οπικισμού. Όσες θυσίες και όσα δεινά και αν χρειαστεί να υποφέρουμε. Γι' αυτό σας ζητώ να μας βοηθήσετε. Είστε φίλοι μας. Βοηθήστε μας να εξαφανιστούν όλα αυτά τα δεινά. Αυτό που γεννάει την απελπισία αυτή και τη ματέωση που ζει ο λαός μας. Έτσι ώστε να μπορέσουμε να τερματίσουμε την πιο μακροχρόνια κατοχή της σύγχρονης ιστορίας. Δεν υπάρχει ε, άλλο τέτοιο παράδειγμα τέτοιας διάρκειας. Βοηθήστε μας να τερματίσουμε την κατοχή αυτή. Ο Παλαιστινιακός λαός είναι από τους αρχαιότερους λαούς του κόσμου και στην περιοχή και παγκοσμίω. Έχουμε από τους παλαιότερους αρχαιότερους πολιτισμούς. Είναι λογικό να στερείται του ίδιου του, του κράτους ο λαός αυτός. Δεν έχει έρθει η ώρα ο λαός μας να μπορέσει επιτέλους να ζει ελεύθερα χωρίς να περνάει checkpoint, ελέγχους, φυλάκια, χωρίς τύχη, χωρίς ε, διαβάσεις και περάσματα που μπορεί να ανοιγοκλίνει κατά το δοκούν και αυθαίρετα ο Ισραηλινός στρατός. Κυρίες και κύριοι, το Ισραήλ έχει κάνει τη χώρα μας μια, υπεύθυα, ε, μια υπαίθρια φυλακή για το λόγο μας. Κυρίες και κύριοι, εδώ ενώπιόν σας θα ήθελα να επαναλάβω ότι εμείς δεν θέλουμε να καταργήσουμε κανένα, ούτε να σβήσουμε κανένα από το γεωγραφικό χάρτη, όπως ορισμένοι ισχυρίζονται. Ούτε μπορεί να καταργήσει κανένα. Ούτε επιθυμούμε κάτι τέτοιο εμείς. Αυτό που θέλουμε είναι να, το δικαίωμα στην ύπαρξη. Αλλά δεν θα επιτρέψουμε επίσης να προσπαθήσει κάποιος να μας σβήσει εμάς. Να σβήσει τη δική μας παρουσία και ύπαρξη από ε, τη γη μας, να σφετεριστεί τα δικαιώματά μας. Η μόνιμη και επίμονη άρνηση ε, το, αναγνώριση των δικαιωμάτων μας εξυπηρετεί μόνο τους εξτρεμιστές και γεννάει τρομοκρατία και βία. Δίνει στους βίους και στους τρομοκράτες και στους ε, ακραίους προφάσεις και δικαιολογίες. Γι' αυτό σας ζητώ να μην επιτρέψετε η, ε, η υπόθεση της Παλαιστίνης να γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης από τους εξτρεμιστές αυτούς. Θα πρέπει όλοι οι εξτρεμιστές αυτοί να σταματήσουν τη δράση αυτή και να ξαναγίνει ε, μοντέλο και υπόδειγμα ε, ελευθερίας, δικαιοσύνης και ισότητας ε, η χώρα μας. Απευθυνόμαστε σε εσά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα θεσμικά σα όργανα, για να συνεχίσετε τι προσπάθειέ σα και τι διπλωματικέ και τι πολιτικέ, έτσι ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια δίκαιη λύση στη περιοχή μα. Και αυτό βάσει τη ε, λύση των δύο κρατών εντό των συνόρων του 1967, όπω είπε ο κύριο Πρόεδρο προηγουμένω, και χάρη στο σεβασμό των διεθνών ψηφισμάτων. Το Ισραήλ και η Παλαιστίνη έχουν δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν και συμφωνίες σύνδεσης μαζί της. Και οι δύο είναι μέλη της Ένωσης ε, για τη Μεσόγειο. Το αποτέλεσμα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί ένα πολύ σημαντικό παίκτη. Από αυτό μπορούν να αποφεληθούν όλες οι πλευρές. Κυρίες και κύριοι, θέλω να σας μιλήσω ειλικρινά έτσι συνηθίζω να μιλάω όταν συνομιλώ με οποιονδήποτε. Και έτσι θα μπορέσω νομίζω να απαντήσω και σε κάποιες απορίες που ίσως έχετε. Εμείς είμαστε υπέρ της λύσης των δύο κρατών. Θέλουμε να δημιουργηθεί το κράτος της Παλαιστίνης σε ολόκληρη την επικράτεια της Δυτικής Όχθης. Στα σύνορα της 4ης Ιουνίου του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ η οποία βρίσκεται υποκατοχή από τότε. Δεν είμαστε κατά του να γίνει κάποια ανταλλαγή εδαφών, υπό τον όρο βέβαια ότι θα είναι ίδιας αξίας και σε ένα βαθμό μόνο. Είναι απαραίτητο να αντιμετωπίσουμε το θέμα των προσφύγων βάσει του ψηφίσματος 194 και βάσει της πρωτοβουλίας η ε, ειρήνης της αραβικής ειρηνευτικής πρωτοβουλίας η οποία ζήτησε μια δίκαια λύση και διαπραγμάτευση όσον αφορά το πρόβλημα των προσφύγων. Αυτή η αραβική πρωτοβουλία αποτελεί και μέρος του χάρτη πορείας. Βάσει του ψηφίσματος 1515 του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και πρέπει να σας πω ότι έχουμε αναγνωρίσει το, ο, η οργάνωση για την Παλαιστίνη το 1993 αναγνώρισε το κράτος του Ισραήλ. Ακριβώς γι' αυτό λοιπόν και εμείς θέλουμε ειρήνη για όλους. Και δεχτήκαμε να υπάρχει ένα τρίτο μέρος στα σύνορά μας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη μελλοντική Παλαιστίνη. Συμφωνήσαμε δηλαδή με μέτρα ασφάλειας περιφερειακού χαρακτήρα. Όμως αρνούμεθα πλήρως τις προσωρινές λύσεις, γιατί είναι χάσιμο χρόνο και τίποτα άλλο. Ούτε δεχόμαστε ένα Παλαιστινιακό κράτος με προσωρινά σύνορα. Επιθυμούμε η Αραβική Ειρηνευτική Πρωτοβουλία, η οποία εγκρίθηκε στη Βηρητό το 2002, αυτή να εφαρμοστεί, να υλοποιηθεί χωρίς καμία τροποποίηση. Οι Ισραηλινοί συχνά αναφέρονται στις ε, κινήσεις ε, προς επιθέσεις, μα αυτές δεν σταματούν από πλευράς του Ισραήλ, γιατί είναι οι έπικοι αυτοί που τους προκαλούν. Για να αποφύγουμε λοιπόν κάθε τέτοια κίνητρα από πλευράς των ακραίων, εμείς θέλουμε η τριμερής επιτροπή Ισραήλ, Παλαιστίνη και Ηνωμένε Πολιτείε να αποκτήσει νέο δυναμισμό. Είναι μια επιτροπή αυτή η οποία δημιουργήθηκε στο White River το 1999 ακριβώς για να λυθούν όλα τα προβλήματα που είχαν να κάνουν με τις βίες πράξεις εκατέρωθεν. Οι Ηνωμένε Πολιτείε αποτελούν το διαιτητή κατά κάποιο τρόπο. Θα λοιπόν υπέρ η Επιτροπή αυτή να αποκτήσει νέο δυναμισμό και η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποτελέσει το τέταρτο μέρος σε αυτό το σχήμα. Αυτό πιστεύω ότι αποτελεί απόδειξη που αποδεικνύει ότι εμεί είμαστε κατά τέτοιων επιθέσεων. Είμαστε κατά οποιασδήποτε τάσεις που οδηγεί στον εξτρεμισμό. Και εμείς θα θέλαμε να υπάρχει και κάποιος διαιτητής ο οποίος να αποφασίζει τελικά ποιος είναι αυτός που υποδαβλίζει την κατάσταση. Το να συνεχίζουμε να λέμε ότι είναι οι Παλαιστίνοι οι οποίοι προκαλούν τη βία είναι κάτι το οποίο δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Και οι Ισραηλινοί κάνουν το ίδιο. Και θα έπρεπε κάποιος να μπορέσει να παίξει αυτό το ρόλο του διαιτητή σε αυτή την υπόθεση. Η σε αυτή επιτροπή και γιατί όχι να μην γίνει τέτραμερή με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσε κάλλιστα να αποκτήσει νέο δυναμισμό και να παίξει αυτό το ρόλο. Θα ήθελα επίση να σα πω ότι κάποιοι ραβίνοι στο Ισραήλ ανακοίνωσαν σαφέστατα, είπανε στην κυβέρνησή του, να δηλητηριάσουν τα ύδατα για να σκοτωθούν οι Παλαιστίνοι. Αυτό τι είναι. Δεν είναι όθηση στη βία. Δεν είναι ξεκάθαρα μια όθηση στο έγκλημα, στη γενοκτονία. Ον κατά τέτοιων ε, δηλώσεων υπέρ της βίας. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας πω εδώ ότι εάν σταματούσε η κατοχή και ο επικισμός, θα μπορούσε να ζήσει κυρίαρχα το Παλαιστινιακό κράτος και αυτό θα μπορούσε να γίνει γρήγορα. Θα μπορούσε να αποτελέσει ένα θετικό στοιχείο το Παλαιστινιακό κράτος. Θα μπορούσαμε να είμαστε ένας παραπάνω παίκτη ποιότητας, μια όαση ειρήνης που όλοι επιθυμούν. Θα μπορούσαμε να είμαστε ένας υπεύθυνο παίκτη. Ένα Παλαιστινιακό κράτος με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμα, μια ανοιχτή πόλη, ανοιχτή σε όλες τις τρεις θρησκείες που κατοικούν εκεί γύρω. Τον Ιδεσμό, τον χριστιανισμό και το Ισλάμ. Η Ιερουσαλήμ θα ήταν μια ανοιχτή πόλη, γιατί εμεί σεβόμαστε τις τρεις αυτές θρησκείες. Και οι θρησκείες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εκφράζονται ελεύθερα στην Ιερουσαλήμ. Μια πόλη που, όπως είπα, πρέπει να παραμείνει ανοιχτή. Η χώρα μας, με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούσε υπεύθυνα να διαχειρίζεται τις υποθέσεις της, την ανάπτυξή της, να διαχειρίζεται τους φυσικούς της σπόρους. Όταν θα έχουμε 60% της επικρατείας μας, θα μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε και τους ανθρώπινους σπόρους καλύτερα. Γιατί τα εδάφια αυτά σήμερα αποτελούν τη ζώνη Γ μετά από την συμφωνία του Όσλο. 60% δηλαδή της επικράτειάς μας είναι κομμάτι με το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Είναι ένα κομμάτι στο οποίο δεν μπορούμε να ασκήσουμε ούτε τη γεωργία, ούτε να έχουμε βιομηχανία, ούτε τίποτα. Είναι μία δηλαδή περιοχή στην κατηγορία Γ, η οποία βρίσκεται υποκατοχή από τον Ισραηλινό στρατό και όπου το Ισραήλ και ο στρατός του φέρουν σε πέρας παράνομα σχέδια. Από το 1996, αν λοιπόν μπορούσαμε να πάρουμε πίσω τα εδάφια αυτά, θα μπορούσαμε να κάνουμε θαύματα στη γεωργία, στη βιομηχανία, στον τουρισμό και αναρωτιέμαι γιατί οι Ισραηλινοί επιμένουν τόσο να παραμένουν εκεί. Θα μπορούσαμε λοιπόν έτσι να αναπτύξουμε προγράμματα βιομηχανικά, αγροτικά και θα μπορούσαμε να δώσουμε και δουλειά σε δεκάδες χιλιάδες νέους. Θα μπορούσαμε να, εκπε... να εκμεταλλευτούμε καλύτερα τους φυσικούς μας πόρους, πετρέλαιο, φυσικό αέριο. Θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε καθαρό ηλεκτρισμό. Έχουμε σχέδια. Έχουμε την κοιλάδα του Ιορδάνη. Έχουμε πολλούς χώρους όπου θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε τέτοια προγράμματα και τουρισμό, γιατί μην ξεχνάτε ότι πολλοί έρχονται να προσκυνήσουν είτε στην Βιθλέμ είτε στην Ανατολική Ιερουσαλήμ αν μας δώσετε κράτος, δεν χρειαζόμαστε καμία βοήθεια. Έχουμε πολλούς, ε, πολλά θετικά, πολλά πλεονεκτήματα, αν έχουμε το κράτος μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας βοήθησε, όπως και άλλες φίλες χώρες. Μας βοηθήσατε να δημιουργήσουμε την αρχή αυτού του κράτους. Θα συνεχίσουμε λοιπόν τις προσπάθειές μας στην οικοδόμηση του Παλαιστινιακού κράτους, γιατί το δίκαιο στην αυτοδιάθεση για τον Παλαιστινιακό λαό δεν εξαρτάται από τις διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ. Το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση δεν υποβάλλεται σε διαπραγματεύσεις. Είναι ένα φυσικό δικαίωμα. Χρειαζόμαστε λοιπόν τη βοήθειά σας. Έχουμε σχολεία, πανεπιστήμια, εκπαιδευτικούς θεσμούς δηλαδή, πολύ υψηλού επίπεδου. Κάτι το οποίο μας επιτρέπει να βελτιώσουμε τους δείχτες στον τομέα του αλφαβητισμού και της εκπαίδευσης. Έχουμε ερευνητικά ιδρύματα επίσης. Μικτά. Είμαστε μια ελεύθερη κοινωνία, όπου η γυναίκα είναι ισότιμη με τον άντρα. Πλήρως, είναι ίση, έχουν τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις και οι δύο. Κυρίες και κύριοι, κύριε Πρόεδρε, στις 3 Ιουνίου μια υπουργική συνάντηση έλαβε χώρα στο Παρίσι μετά από γαλλική πρωτοβουλία. Και εκεί συμμετείχαν 28 χώρες και τρεις διεθνείς οργανισμοί. Ευχαριστούμε πολύ για αυτήν την ευγενή προσπάθεια που έγινε και αυτή η πρώτη προσπάθεια καλό θα ήταν να δώσει συνέχεια και να καταλήξει σε μια διεθνή διάσκεψη για το διεθνές δίκαιο και την διεθνή νομιμότητα βάσει των ψηφισμάτων που ισχύουν του Συμβουλίου Ασφαλείας και βάσει της Αραβικής Ειρηνευτικής Πρωτοβουλίας που εγκρίθηκε το 2002 στη Βηρητό και βάση και του χάρτη πορείας όλων των άλλων συμφωνιών που έχουν υπογραφεί. Θα έπρεπε, εάν και εφόσον λάβει χώρα η διάσκεψη αυτή, θα έπρεπε να επιβληθούν και προθεσμίες. Δεν είναι δυνατόν οι διαπραγματεύσεις να γίνονται πάπυρο, ισαΐ, χωρίς να καταλήγουν. Οι διαπραγματεύσεις είναι σημαντικές, αλλά η εφαρμογή των συμφωνιών και αυτή πρέπει να υποβάλλεται σε προθεσμίες. Θα ήταν καλό λοιπόν να δημιουργήσουμε έναν μηχανισμό παρακολούθησης των συμφωνιών αυτών, όπως ακριβώς έγινε και με το Ιράν. Η ομάδα 5 συν 1 στην περίπτωση του Ιράνα επέτρεψε ακριβώς να λυθεί το πρόβλημα και θα ήταν καλό να έχουμε έναν αντίστοιχο μηχανισμό 7 συν 2 ή όποιος μηχανισμός και αν είναι να είναι ένας μηχανισμός παρακολούθησης των αποτελεσμάτων της διάσκεψης αυτής που επιθυμώ να λάβει η χώρα κάποια στιγμή. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει εγκρίνει στην τελευταία του συνεδρίαση ένα τελικό ανακοινωθέν ε, σε σχέση με τη συνδιάσκεψη που έγινε στις 3 Ιουνίου το Παρίσι, εμείς και οι Άραβες αδελφοί μας υποστηρίζουμε τη γαλλική πρωτοβουλία. Ο κύριος Φρανσουά Ολάντο, πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, μου είπε πριν από λίγες μέρες ότι η Γαλλία είναι αποφασισμένη να συνεχίσει τις προσπάθειές της ώστε μια διεθνής συνδιάσκεψη ειρήνης να μπορέσει να λάβει χώρα πριν από το τέλος του 2016. Αναφέρθηκε στην ανάγκη να ξεκινήσουν οι προπαρασκευαστικές εργασίες για μια τέτοια συνδιάσκεψη ώστε να εξασφαλίσουν και την επιτυχία της. Οι ομάδες εργασίας και οι λεγόμενοι ΣΕΡΠΑ θα πρέπει να προετοιμάσουν τις ε, εργασίες αυτές της συνδιασκέψεως. Εγώ ως Παλαιστίνιος, ως Άραβας, είμαι μαζί σας για να γίνει αυτός ο αγώνας εναντίον της τρομοκρατίας και του, και του εξτρεμισμού. Βρισκόμαστε στο ίδιο χαράκωμα. Όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή είναι τα ίδια τα οποία σημαίνουν και στην Ευρώπη, στις Βρυξέλλες, στο Παρίσι, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είμαστε όλοι αντίπαλοι της τρομοκρατίας ανεξάρτητα με τη μορφή που που παίρνει η τρομοκρατία και ανεξάρτητα από τους δράστες αυτών των τρομοκρατικών ενεργειών. Είμαστε στεναρά κατά της τρομοκρατίας. Για να μπορέσουμε όμως να μπορέσουμε να υπερνικήσουμε την τρομοκρατία θα πρέπει να θέσουμε τέμπλωμα και στην κατοχή της Παλαιστίνης από το Ισραήλ. Με το να δημιουργηθεί ένα Παλαιστινιακό κράτος στα όρια του 1967 με την Ανατολική Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα. Μόνο έτσι θα μπορέσουν οι Παλαιστίνοι να ζήσουν σε ειρήνη και ασφάλεια πλάι-πλάι με τους Ισραηλινούς. Χωρίς μια τέτοια λύση δεν θα μπορέσει να ξεπεραστεί η τρομοκρατία θα δίνουμε πάντα όπλα και προσχήματα στους τρομοκράτες οι οποίοι φωνεύουν στο όνομα της θρησκείας. Από τη στιγμή λοιπόν που θα έχει περατωθεί αυτή η κατοχή δεν θα υπάρχουν πλέον τέτοια προσχήματα και ο εξτρεμισμός θα έχει υπερνικηθεί και η τρομοκρατία. Δεν θα υπάρξει πια τρομοκρατία ούτε στη Μέση Ανατολή ούτε στον υπόλοιπο κόσμο. Η αρχή λοιπόν της λύσης του προβλήματος της τρομοκρατίας ξεκινά από την Παλαιστίνη κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Η μη ύπαρξη ενός Παλαιστινιακού κράτους <clears throat> οδηγεί στη διαώνιση της αντιπαράθεσης στη Μέση Ανατολή. Αυτό εξυπηρετεί μοναχά τα συμφέροντα των τρομοκρατών, των εξτρεμιστών, αυτών που θέλουν τη βία. Πολλές χώρες έχουν πληγεί από αυτή τη βία και στη δική μας περιοχή και ευρύτερα είναι θύματα μιας τρομοκρατίας που οδήγησε σε μεγάλα κύματα προσφυγιάς και οδήγησε τους πρόσφυγες αυτούς που φτάνουν στην Ευρώπη σήμερα. Υπήρξαν Παλαιστίνοι πρόσφυγες που υπήρξαν θύματα αυτής της κατάστασης. Σας ζητούμε να αντιμετωπίσετε και τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες όπως και όλους τους άλλους πρόσφυγες σήμερα γιατί χρειάστηκε να φύγουν από τις αιστείες τους για να γλιτώσουν από τον πόλεμο τις φαγές και μια τρομοκρατία την οποία καταδικάζουμε απερίφραστα. Η τρομοκρατία είναι αυτή που οδηγεί στα μεγάλα κύματα προσφύγων. Μεταξύ αυτών των προσφύγων όμως υπάρχουν και οι Παλαιστίνοι πρόσφυγες. Εμείς δεν έχουμε ξεκινήσει λόγω εσωτερικών συγκρούσεων στην περιοχή μας. Αλλά είμαστε αυτοί οι οποίοι έχουμε πληρώσει το τίμημα αυτών των συγκρούσεων. Και παρόλα αυτά, εμείς δεν έχουμε το δικαίωμα ως Παλαιστίνοι πρόσφυγες τα ίδια δικαιώματα που έχουν οι άλλοι πρόσφυγες στον κόσμο. Γιατί λοιπόν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Πρέπει να αλλάξετε την αντιμετώπιση σα. Ο Παλαιστίνιος πρόσφυγα είναι στην ίδια κατάσταση με του άλλου πρόσφυγε. Χρειάζεται συμπόνια, χρειάζεται βοήθεια, χρειάζεται υποστήριξη. <clears throat> Σε ό,τι αφορά τώρα την εσωτερική κατάσταση στην Παλαιστίνη. Θα ήθελα να σας πω ότι εμεί προσπαθούμε να ενώσουμε τα εδάφη μα, να ξεπεράσουμε τον αποκλεισμό ο οποίος πλήττει τη λωρίδα της Γάζας. Προσπαθούμε να ξεπεράσουμε τις εσωτερικές διαμάχες μεταξύ μας με τη δημιουργία μιας κυβέρνησης εθνικής ενότητας η οποία θα σέβεται την πολιτική γραμμή της ε, οργάνωσης για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης και τις διεθνείς και περιφερειακές δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει. Εάν θέλουμε να υπάρξει μια κυβέρνηση για όλη την Παλαιστίνη με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων μερών. Μια κυβέρνηση λοιπόν εθνικής ενότητας. Η κυβέρνηση αυτή θα πρέπει, όπως και όλες οι συνιστώσεις της, να σέβονται αυτές τις δεσμεύσεις. Δεν μπορεί ένα κόμμα να πει ότι δεν θέλει να δεχτεί κάποια από αυτές τις δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει ως Παλαιστίνη. Είμαστε έτοιμοι λοιπόν να προχωρήσουμε σε αυτή την κυβέρνηση εθνική Ενότητα, μετά από την οποία συγκρότηση μπορούμε να περάσουμε σε βουλευτικές και μετά προεδρικές εκλογές για να ξεπεράσουμε το τωρινό καθεστώς διχασμού στα παλαιστινιακά εδάφη. Θέλω να χρησιμοποιήσω την ευκαιρία για να ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλα τα κράτη-μέλη για τις προσπάθειες που έχουν καταβάλει για τη συμβολή τους υπέρ της ανοικοδόμησης αυτών που έχει καταστρέψει στη Γάζα η Ισραηλινή κατοχή. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι έχουν εξαπολυθεί τρεις πόλεμοι κατά της Λόριδας της Γάζας. Είναι χιλιάδες τα θύματα, είναι εκατοντάδες χιλιάδες οι τραυματισμένοι και πάρα πολλά τα εγκύματα και οι εγκαταστάσεις και υποδομές που έχουν καταστραφεί. Αξίζεται λοιπόν την απόλυτη ευγνωμοσύνη μας για τη βοήθεια που μας δώσετε για την ανοικοδόμηση. Κύριε Πρόεδρε, σας ζητώ να ε, δεχτείτε την ευγνωμοσύνη μου γιατί έχω και την ευκαιρία μέσω, πάνω, μέσα από αυτό το βήμα να ε, εκφράσω ένα μήνυμα προς την Ισραηλινή κυβέρνηση. Έχουμε απλώσει χείρα ειρήνης προς σας έχουμε την πολιτική θέληση για να επιτύχουμε αυτή την ειρήνη. Σας ζητώ λοιπόν να απαντήσετε ως Ισραηλινή κυβέρνηση. Έχετε και εσείς την διαθέληση, Είσαστε έτοιμοι να αναθεωρήσετε τη θέση σας και να αναγνωρίσετε την ιστορική αδικία που έχει πράξει η δική σας πλευρά και που έχει κάνει τη δική μας πλευρά να υποστεί. Έχουμε τη δική μας ιστορία, έχετε και εσείς τη δική σας ιστορία. Έχουμε το αφήγημα αυτό το οποίο είναι ειλικρινές. Είναι έντιμο. Η ύπαρξή μας σε αυτά τα εδάφη είναι συνεχής από την αυγή της ιστορίας μέχρι σήμερα. Έχουμε και εμείς σταθερά δικαιώματα για αυτά τα εδάφη και για τους ιερούς μας τόπους, είτε είναι χριστιανικοί είτε είναι εβραϊκή είτε μουσουλμανική. Η ειρήνη και η συμφιλίωση δεν μπορούν παρά να περάσουν μόνο μέσα από την αναγνώριση των δικαιωμάτων μας και την αποζημίωση για τις καταστροφές. Κανείς δεν έχει συμφέρον να μεταμορφώσει ένα πολιτικό αγώνα σε μια θρησκευτική αντιπαράθεση. Αυτό θα ήταν ένα πραγματικό κίνδυνο. Αυτή η διαμάχη λοιπόν δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι είναι σύγκρουση θρησκειών. Θα πρέπει τα θρησκευτικά θέματα να αφαιθούν κατά μέρο. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια πολιτική αντιπαράθεση. Οποιαδήποτε λύση δεν μπορεί να είναι παρά μόνο πολιτική. Το να χρησιμοποιήσει κανεί θρησκευτικά προσχήματα αυτό οδηγεί σε πραγματικούς κινδύνους, σε πραγματικές απειλές για όλους μας. Όλοι έχουν συμφέρον να επικρατήσει η ειρήνη. Ελπίζω ότι εσείς, οι γειτονέ μας, οι Ισραηλοί και εσείς πιστεύετε στην ειρήνη. Ας οικοδομήσουμε λοιπόν την ειρήνη. Ας οικοδομήσουμε μια ειρήνη πέραν της ηγεμονίας της απικιοκρατίας και των επικισμών. Μια ειρήνη η οποία να βασίζεται στη συνύπαρξη, στο κράτος δικαίου, του αμοιβαίου σεβασμού και του σεβασμού της αξιοπρέπειας και της ελευθερίας όλων στην περιοχή μας. Μόνο μια τέτοια ειρήνη μπορεί να αποτελέσει τον πραγματικό εγγυητή για τη σταθερότητα, για την ειρήνη και για ένα ελπιδοφόρο μέλλον για τις επερχόμενες γενιές. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ και πάλι για την υποδοχή σας και θέλω να σας πω ότι βασιζόμαστε στις ευγενείς προσπάθειές σας για να επανέλθει η ειρήνη στην περιοχή μας. Ζήτω η ευρωπαλαιστινιακή φιλία. Ας γίνει η γη της Παλαιστίνης, η οι Άγιοι τόποι ας γίνουν μια όαση ειρήνης και σταθερότητας και για τον Παλαιστινιακό λαό και για τους γείτονές του και για όλο μας τον κόσμο. Σήμερα έχουμε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για αυτά τα οποία λαμβάνουν χώρα στη Μεγάλη Βρετανία και παρακολουθούμε από πολύ κοντά τα τεκτενόμενα. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να ευχαριστήσω τον πρόεδρο μα. Σα ευχαριστώ για τα λόγια σα. Χθε ήταν παρόν ο πρόεδρο του Ισραήλ, ο οποίο ομίλησε και στα αραβικά. Θα ήθελα και του ε, δύο από εσά να σα ενθαρρύνω να καθίσετε στην τράπεζα του διαλόγου και των διαπραγματεύσεων και εμεί θα υποστηρίξουμε απόλυτα τι προσπάθειε σα. Ευχαριστώ. Wznawiam posiedzenie. Witam bardzo. Συνεχίζουμε τη συνεδρίαση και σας καλωσορίζω όλους. Παρακαλώ. Θα ψηφίσουμε. Καλωσορίζω τους βουλευτές του Κρανικού Κοινοβουλίου και τον πρόεδρο της Ουκρανικής Διαστημικής Υπηρεσίας. Και περνάμε τώρα